έχει δημοσιευθεί ε, και στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η αυριανή ημερήσια διάταξη και θα ήθελα εδώ να διακόψουμε και να ευχηθώ σε όλους σας ε, καλό